δικά της τρέχουσας συνεδρίασης. Και προχωρώ στην ημερήσια διάταξη και τις αλλαγές της, ή καλύτερα την έγκρισή της, δυνάμει του άρθρου 137, ελήφθη απόφαση από το Προεδρείο, από τη των Προέδρων για την έγκριση για τον προσορισμό της ημερήσια διάταξης στις 7 Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ορίζεται η ημερήσια διάταξη για την τρέχουσα σύνοδο.